Όχι, ωραία, εγκρίνονται. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Ιζαμπέλα Λεβίν από 3 Οκτωβρίου ε, ορίστηκε Υπουργός Ανάπτυξης της Σουηδίας και την συγχαίρω. Οι, οι αρμόδιες ε, ελβετικές αρχές ε, με ενημέρωσαν πως αντικαθίσταται από την κυρία Λινέα Έγκστρομ από 8 Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγραφός 1 του κανονισμού όπως επίσης και με βάση το άρθρο 4 παραγραφός 1 και 4 θεωρεί πως είναι βουλευτής η κυρία Λινέα Έγκστρομ από τις 8 Οκτωβρίου 2014 και υπενθυμίζω πως σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 κάθε βουλευτής συμμετέχει στις επιτροπές της εργασίες του Κοινοβουλίου μέχρι να διαπιστωθεί πως έχει προσκομίσει σωστά τα ε, τα διαπιστευτήριά του ή μέχρι να υπάρξει κάποια αντίρρηση. Ο κύριος Γιώχαν Φαν Όβερφελτ από 11 Οκτωβρίου 2014 έγινε Υπουργός Οικονομικών του Βελγίου. Συγχαίρω τον κύριο Φαν Φαν-Οβερτφέλτ και βεβαίως σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού θεωρούμε πως η θέση αυτή χειρεύει και πρέπει να πληρωθεί. Ο κύριος Ρίχαρτ Ζούλικ έφυγε από την ομάδα Άλντε και πήγε στην ομάδα ECR από τις 8 Οκτωβρίου 2014. Από την Γκουε, ε, Άλντε,